Hello. Uh, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις για να αρχίσουμε αμέσως τη συνεδρίασή μας. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu Αρχίζει και πάλι η συνεδρίασή μας που διεκόπη στις 9 Σεπτεμβρίου του 2010. Και με μεγάλη λύπη μου πρέπει να σας ανακοινώσω τον θάνατο του Έγκον Κλέψου που ήταν